συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ε, ψηφοφορία αύριο στις 12. Η... Δημοσιεύτηκε η αυριανή ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια. Σας εύχομαι και σας